Mes chers collègues, je Άρχεται η συνεδρίαση. Η συνεδρίαση της ΕΚΟΝ και των προϋπολογισμών. Θα ήθελα τη σύμφωνη γνώμη σας για την ημερήσια διάταξη. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θεωρώ ότι εγκρίνεται. Και θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι υπήρχε συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ΕΤΕ για την ανταλλαγή πληροφοριών μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας του ΕΦΣΥ. Όπως ξέρετε έγινε πληθώρα συζητήσεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και το θέμα ε, και θα υποβληθεί στη διάσκεψη των Προέδρων και θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο τον κύριο Ταγιάννη. Και θα είναι στη διάθεσή σας αν δεν έχει ήδη γίνει. Περιμένουμε τους δύο εισηγητές μας, τους Φερνάντες και Μπούλμαν, για να αποτιμήσουν την κατάσταση του ΕΦΣΥ. Έχουν στη διάθεσή τους 10 λεπτά και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στους κοιόδης για 2 λεπτά τον καθένα. Στη συνέχεια θα ακούσουμε και ε, τους εκπροσώπους της ΕΤΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε πολύ φορτωμένη ημερήσια διάταξη γιατί πρέπει ανυπερθέτως να τελειώσουμε στις 19.50 έτσι ώστε να ψηφίσουμε στις 8 παρα την έκθεση Μπέρες σε σχέση με την δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης και στις 8 η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων θα ασχοληθεί με άλλα ζητήματα μαζί με την Επιτροπή Προϋπολογισμό. Δίνω το λόγο στον κύριο Μπούλμαν για πέντε λεπτά. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες με τον οποίο ε, συνυποβάλλω αυτή την έκθεση προς εξέταση. Αγαπητοί μου συνάδελφοι, πράγματι πιστεύουμε ότι κάναμε καλή νομοθετική δουλειά και ταχεία νομοθετική δουλειά για να μπει σε πρόγραμμα το ΕΦΣΥ. Η νομοθεσία ανέδειξε κάποια θέματα, ζητάει γνήσια προσθετικότητα, ενίσχυσε τις ε, διάμεσες δομές, ε, θέλει να πάρουν κεντρικό ρόλο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αυτά τα project. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την νομοθεσία, αλλά όχι πάντα, το λέω ευθύς εξ αρχής, όχι πάντα ε, με τον τρόπο της υλοποίησης. Φαίνεται ότι η ποσοτική στόχη ε, εφαρμόζονται αλλά υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες εις ό,τι αφορά την ποιότητα. Οι ποσοτικοί στόχοι εφαρμόζονται, αλλά η ποιότητα των project καμιά φορά ε, δημιουργούν πρόβλημα. Η προσθετικότητα είναι ένα ερωτηματικό, αν ε, είναι όλα τα project προσθετικά. Έκλεισε το μικρόφωνο. Τώρα ακούγεται. Υπάρχουν αμφιβολίες εις ό,τι αφορά την βιώσιμη υλοποίηση των διατάξεων της νομοθεσίας στην χρήση του scoreboard, για παράδειγμα, του πίνακα επιδόσεων που επανυπέβαλε το Κοινοβούλιο. Η Τράπεζα Επενδύσεων αναφέρει στην ετήσια έκθεση ότι αυτό το scoreboard ε, μπαίνει, θα πρέπει να μετράει και τους νέους ε, πυλώνες αλλά όχι να χρησιμοποιείται για την ε, διάρθρωση και ιεράρχηση των έργων. Επίσης ο έλεγχος των project δεν μπορεί να διαρκεί τόσο πολύ ώστε οι υποβάλλοντες στο έργο να μην ξέρουν τι τους περιμένει ούτε επιτρέπεται ένα κεντρικό μέσο όπως οι επενδυτικές πλατφόρμες να τις χρησιμοποιούμε ε, ε, να μην τις χρησιμοποιούμε ή να τις χρησιμοποιούμε λίγο ενώ ε, έχουν συσταθεί για την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων. Βλέπουμε μια σύγκρουση μεταξύ του ποσοτικού στόχου και της ποιότητας των έργων, των projects. Ενδεχομένως θα έπρεπε να μιλήσουμε και με τους υπεύθυνους από την Τράπεζα Επενδύσεων και το ΕΦΣΙ για να αποφευθούν συγκρούσεις και να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ των ε, ποιοτικών στόχων και των καινοτόμων ε, στόχων των projects. Αυτά όλα πρέπει να τα δούμε πριν περάσουμε στη νομοθέτηση του ΕΦΣΙ 2. Πρέπει να προσέξουμε ώστε η γεωγραφική κατανομή των επενδύσεων να είναι σωστή και τα κονδύλια να φτάνουν εκεί που χρειάζονται περισσότερες πρόσθετες επενδύσεις, γιατί και αυτό δεν είναι πάντα ξεκάθαρο. Θέλουμε περισσότερη διαφάνεια, είναι προφανές αυτό στα πλαίσια της πρότασής μας και θέλουμε να δούμε αν η δομή διακυβέρνησης εφαρμόζεται όπως έχει εκλεγεί. Θεωρούμε ότι αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη. Υπάρχει πολλή αδιαφάνεια ακόμη, πολλά ερωτηματικά αμφισβητήσεις στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν. Και η έκθεσή μας αξιολόγησης αυτό θέλει να προκαλέσει μια κριτική ε, αντιπαράθεση και συζήτηση. Ξέρω ότι ο συνάδελφος Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες εστιάζει ιδιαίτερα στην εφαρμογή στις περιφέρειες αυτό τον ενδιαφέρει όλος ιδιαιτέρως διότι επιθυμεί η υποστηρικτική υποδομή να μην υπολείπεται, να είναι στη θέση της σωστής γιατί χρειαζόμαστε μια νέα ικανότητα outreach προβολής αυτών των έργων. Θα τα πει ε, σε λίγο και θα τονίσει αυτό το θέμα. Οπότε δεν συνεχίζω εγώ πάνω σε αυτό. Να προσθέσω ακόμη ότι κάναμε ένα workshop με ειδικού εμπειρογνώμονες που μας ε, βοήθησαν πολύ την προηγούμενη εβδομάδα και θα συμπεριλάβουμε αυτά που μας είπαν και με τη μορφή τροπολογιών και θα τα πούμε και στη συζήτηση που θα ακολουθήσει τώρα συνάδελφοι. Ε, χαιρόμαστε πολύ για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Η ε, προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 28 Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Μπούλμα. Ο Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντες έχει το λόγο από την Επιτροπή των Προϋπολογισμών. Ευχαριστώ. Ε, πρόεδρε, θα μιλήσω πορτογαλικά. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπούλμαν για την εργασία του, την εργασία μας σε σχέση με τα επενδυτικά σχέδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα πλαίσια αναπτυξιακών και εργασιακών προγραμμάτων. Το σχέδιο Juncker ή μάλλον καλύτερα το ΕΦΣΙ περιλαμβάνει το σχέδιο Juncker. Μιλάμε για 168 δις σε 28 κράτη-μέλη και όσον αφορά τις ΜΜΕ, δηλαδή ε, επιχειρήσεις μέχρι, που απασχολούν μέχρι 3.000 εργαζόμενους, συμπεριλαμβάνονται και αποτελούν το επίκεντρο του ΕΦΣΥ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Αν και δεν μπορούμε πάντα να ποσοστοποιήσουμε τους στόχους, όμως σε αυτή την περίπτωση λαμβάνουμε υπόψη της ΜΜΕ όπως αρχικά προβλεπόταν. Υπάρχουν ελλείψεις ως προς τα επενδυτικά προγράμματα, το οποίο σημαίνει ότι αυτό το μέσο θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, για τις επενδύσεις, αλλά και για την αλλαγή προσέγγισης του ΕΤΕ ως προς τις πλατφόρμες που θα χρησιμοποιήσουμε και θα δημιουργήσουμε μεταξύ κρατών μελών, έτσι ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία. Υπάρχουν βελτιώσεις, αλλά και περιθώρια περαιτέρω βελτιώσεων. Ας μιλήσουμε για την προσθετικότητα που είναι μία αμφίσιμη έννοια. Λέμε ότι είναι δύσκολο να ορίσουμε καλύτερα την προσθετικότητα από τον ορισμό που έχουμε. Όμως η ΕΤΕ θα πρέπει να ερνεύσει το γράμμα και το πνεύμα του κανονισμού. Μιλάμε και για ε, εμπροστοβαρείς επενδύσεις με βάση την αρχή της προσθετικότητας. Και γιατί κάτι ή πώς θεωρείται προσθετικό, πώς έχει προσθετικό χαρακτήρα. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει και από πλευράς διαφάνειας. Άρα τα προγράμματα που εγκρίνονται θα πρέπει να δικαιολογούνται πλήρως, να αιτιολογούνται πλήρως. Και το ίδιο ισχύει και για τα προγράμματα που απορρίπτονται. Σε σχέση τώρα με τις πλατφόρμες επενδύσεων σχετίζονται και με μικρότερα προγράμματα ή διασύνοριακά προγράμματα για την εκτέλεση των σχεδίων της αγοράς ενέργειας ιδιαίτερα. Πέρα από αυτό, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την επιτόπια κατάσταση. Δηλαδή άλλο 50 εκατομμύρια ευρώ στο Βερολίνο και άλλο το αντίστοιχο ποσό στην Πορτογαλία. Και επίσης και μέσα στην Πορτογαλία υπάρχουν διαφορές, δηλαδή άλλο 50 εκατομμύρια στο νότο της Πορτογαλίας και άλλο στο βορρά. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη και την εδαφική ε, ακαιρεότητα. Και φυσικά χρειαζόμαστε και αυτή την πλατφόρμα χορήγησης συμβουλών έτσι ώστε να υπάρξει μία αναδιάρθρωση εκεί που θα χρειαστεί. Και επιμένω σε αυτή την πλατφόρμα χορήγηση συμβουλών, πλατφόρμα συμβουλών δηλαδή, και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την εδαφική ολοκλήρωση και ακεραιότητα. Πρόκειται για ένα ανοιχτό ταμείο το οποίο πέρα από τη διαφορετικότητα των τομέων λαμβάνει υπόψη και την εδαφική διαφορετικότητα. Δηλαδή δεν υπάρχει γεωγραφικός συγκεντρωτισμός. Γι' αυτό θέλουμε αυτή την συμβουλευτική πλατφόρμα για να λάβει υπόψη την περιφερειακή πραγματικότητα. Και έτσι ώστε να μην αποκλειστούν επενδύσεις Επίσης, τα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής και επενδύσεων θα μπορούσαν να λάβουν κονδύλια και από το ΕΦΣΥ. Αλλά το ΕΦΣΥ δεν θα αντικαταστήσει την πολιτική συνοχής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τους δύο εισηγητές που μας ε, σκιαγράφησαν την κατάσταση και τα περιθώρια εξέλιξης έτσι ώστε το εύση να γίνει πιο αποδοτικό. Τώρα το λόγο έχουν οι σκιώδεις, δύο λεπτά ο καθένας και θα ήθελα να τηρήσετε το χρόνο σας. Ο κύριος Κάρας έχει το λόγο, αλλά ο κύριος Σαχάιες θα λάβει το λόγο εξ του. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς ο συνάδελφο μου ο κύριος Κάρας ε, δεν μπορούσε να παραστεί σήμερα το βράδυ και ως σκιώδη ηγητή ε, του ΕΛΚ ε, για το θέμα αυτό στην Αρμόδια Επιτροπή μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω. Και θέλει να υπογραμμίσει ο κύριος Κάρας ότι αυτή η αξιολόγηση του ΕΦΣΥ είναι σημαντική και πρέπει να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για να τρέξουμε στο παρελθόν το ότι επιτύχαμε για 1,5 περίπου χρόνο, αλλά και για το τι πρέπει να γίνει κατά τον επόμενο 1,5 χρόνο. Και αν θέλουμε πράγματι να πετύχουμε, δηλαδή να υπάρξουν επενδύσεις, ποιοτικέ επενδύσεις για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, να γίνουν αλλαγές ε, στο καταστατικό που διέπει το ΕΦΣΥ, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το μέγιστο δυνατό δυναμικό που μπορεί να προσφέρει το πρόγραμμα ΕΦΣΥ. Ο κύριος Κάρας χαιρετίζει την έκθεση η οποία προσφέρει μια πολύ καλή ισορροπία ανάμεσα στα υπέρ και τα κατά που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του ΕΦΣΥ το, τους περασμένους ε, 16-19 μήνες. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, θα προκύψουν και κάποια άλλα κατά την αξιολόγηση. Αυτό το λέει και η Κομισιόν και η ΕΤΕ ε, και ανεξάρτητη σύμβουλη, αλλά και η, το αναφέρει και η γνωμοδότηση της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών. Θέλει να αναφερθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος. Καταρχήν πρέπει να ορίσουμε το πώς ορίζεται η προσθετικότητα στα προγράμματα υψηλού κινδύνου. Μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής στον πίνακα επιδόσεων. Θεωρεί ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε πλήρως το δυναμικό που προσφέρει αυτή η πλατφόρμα επενδύσεων. Επίσης δέχεται το να υπάρξουν βελτιώσεις όσον αφορά στη συνεργασία με επενδυτικές τράπεζες και κάτι άλλο όσον αφορά τις ε, μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις. Ε, εκεί πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία και αναφέρεται στην επέκταση των εγγύσεων και σε τρίτες χώρες. τάσετε υπέρ του μεγαλύτερου, της μεγαλύτερης χρήσης του ΕΦΣΥ. Αυτά λοιπόν τα θέματα θα τεθούν κατά τους επόμενους μήνες και ο κύριος Κάρας επιθυμεί να ευχαριστήσει όλους τους συναδέλφους για αυτή την έκθεση η οποία αποτελεί μια πολύ καλή βάση για τις επερχόμενες συζητήσεις. Η κυρία Γκαρσία Ζαμπάλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αφού έλαβαν το λόγο οι δύο εισηγητές, δεν έχουμε και πολλά να πούμε. Νομίζω ότι η πρόταση Μπούλμαν Φερνάντες φύγει πολύ σωστά όλα τα ζητήματα που θα πρέπει να μελετήσουμε και να βελτιώσουμε για την προετοιμασία του ε, Σχεδίου Στρατηγικών Επενδύσεων του ΕΦΣΙ. Βεβαίως, ε, τα στοιχεία, τα αριθμητικά στοιχεία είναι πολύ σημαντικά και ε, όπως ελέγχθη δεν πρέπει να δούμε μόνο το ποσοτικό στοιχείο αλλά και το ποιοτικό. Για να σας απαριθμίσω τα θέματα, η προσθετικότητα είναι κάτι που θα πρέπει να εξετάσουμε εις βάθος. Το Κοινοβούλιο έβαλε μεγάλο, έθεσε μεγάλο βάρος στο θέμα της προσθετικότητας. Ήδη προϋπήρχαν προγράμματα επιδοτήσεων και βοηθείας, αλλά θα πρέπει να δούμε μέσα στα πλαίσια του ΕΦΣΥ κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε ένα επιπρόσθετο ποιοτικό βήμα. Για να μην υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την προσθετικότητα, θα πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται και η προεπιλογή που γίνεται πριν φτάσουμε στο τελικό στάδιο επιλογής για να δούμε τι κριτήρια πληρούν αυτά τα προγράμματα, γιατί πολλές φορές δεν έχουμε τις κατάλληλες πληροφορίες ως προς την γεωγραφική κάλυψη. Είναι ένα θέμα που θα πρέπει να εξετάσουμε για να αποζητήσουμε μία εξισορρόπηση και μία γενική αποτίμηση γιατί πολλές φορές κανείς δεν ξέρει καν πώς πρέπει να προβεί στη σύσταση ενός προγράμματος για να είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να βελτιώσουμε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας. Σάντερ Λούνες. Ο συνάδελφός μου θα λάβει το λόγο. Θα μιλήσει εξ του κυρίου Λούνες. Έχετε το λόγο. Να μιλήσω είμαι ε, σκιώδης από το ECR στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Ευχαριστώ τους εισηγητές για το έργο τους. Χαίρομαι Ήδη ε, διαμορφώνεται μια συνένεση στην έκθεση. Πολύ σημαντική είναι η γεωγραφική ανισοκατανομή των επενδύσεων εύση. Από την να ακούμε πόση επιτυχία έχει το εύση. Όμως πρέπει να είναι ειλικρινείς και να πούνε ότι τη μερίδα του Λέοντος την πήραν τα 15 κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης πήραν πολύ μικρά κομμάτια της πίτας. Σημαντικό είναι να συμβάλλει το ΕΦΣΙ στην οικονομική και κοινωνική συνοχή της Ευρώπης στο ε, δεν, θα επαναλάβω τα της προσθετικότητας, συμφωνώ με τις ανησυχίες που εκφράστηκαν. Να προσθέσω κάτι καινούριο όμως, μια καινούρια φωνή που ε, έρχεται από τη διαδικασία έγκρισης των έργων. Προσπαθούν να συνεργαστούν με πολλούς δήμους, με ΟΤΑ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και να ανεβρεθούν ιδιώτες ε, επενδυτές που όμως στην πραγματικότητα ε, είναι δημόσιοι γιατί ε, είναι τα χρήματα των δήμων. σε τελευταία ανάλυση δηλαδή όλα αυτά πληρώνονται από τους φορολογουμένους. Αυτά πρέπει να μας ανησυχούν γιατί ε, πολλές φορές ε, υπάρχουν πολιτικές ε, επιδιώξεις και αυτά δημιουργούν ανισορροπίες και αρνητικό αντίχτυπο ενδεχομένω όλου του Ταμείου Εύση. Αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Ο Ρίτσαρντ έχει το λόγο. Εγώ θα εκπροσωπήσω τον Ρίτσαρντ Έσουαρθ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, να ευχαριστήσω θερμά τους δυο εισηγητές, ε, τους συναδέλφους Φερνάντες και Μπούλμαν για την έκθεση αυτή για την οποία πιστεύω ότι θέτει τις σωστές ερωτήσεις και τα σωστά θέματα. Ε, πράγματι συμφωνώ, πρέπει να εξετάσουμε κριτικά το εύση Αφού τρέχει το έργο, θα κάθε έργο θα πρέπει να ε, ε, έχει τη μεγαλύτερη επιτυχία. Γενικά ε, ε, βλέπουμε όμως ε, να προβάλλονται υπερβολικά τα θετικά. Γιατί εγώ βλέπω κάποια προβλήματα στο ΕΦΣΙ, ότι δηλαδή εδώ προσπαθούμε να καθοδηγήσουμε μέσα από κρατικά μέσα και μηχανισμούς στην αγορά και αυτό είναι λάθος. Και όταν διαπιστώνουμε επενδυτικό κενό και λίγες επενδύσεις στην Ευρώπη, Σωστό είναι να επέμβουμε, αλλά δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε με κρατικές παρεμβάσεις στην αγορά. Διότι έτσι μπορεί να ανάψει μια φωτιά η οποία μπορεί να στοιχήσει πάρα πολύ. Ε, θα δαπανηθούν δηλαδή πολλά κονδύλια και δεν θα έχουν δημιουργηθεί οι σωστές δομές. Αυτή, αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος με το εύση ότι δηλαδή θα δημιουργήσουμε ε, σφάλματα επενδύοντας σε τομείς για τους οποίους δεν ξέρουμε αν θα είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα στην αγορά. Καλύτερα να καταπολεμήσουμε τα αίτια της κρίσης που πού θα τα αναζητήσουμε ε, ε, στην υπερχρέωση κάποιων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιες οικονομίες δεν είναι πια ανταγωνιστικές και αυτό έχει να κάνει με το ευρώ και όχι με την έλλειψη των επενδύσεων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τρεμόζα, τον οποίο δεν βλέπω, ο Νίλ Τόρβαλς έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ε, λέγοντας τα εξής. Έχοντας ακούσει τους δύο εισηγητές και έχοντας διαβάσει την έκθεση, προσβλέπω στη συζήτηση για αυτό το ψήφισμα, αλλά και για την αναθεώρηση γενικά του ΕΦΣΥ. Με ανησυχεί το ότι οι χώρες ε, της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης έχουν πάρει μόνο το 9% των κονδυλίων. Κάτι δεν πάει καλά με αυτό τον αριθμό. Επίσης, ε, αυτή τη στιγμή το ΕΠΣΑ δεν επηρεάζει ουσιαστικά ε, την, ε, τα δίκτυα, τα διευρωπαϊκά, ούτε αυτά που αφορούν στην ενέργεια. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε να εφαρμόζονται, να εκτελούνται περισσότερα προγράμματα υπερεθνικά και να προσφέρουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Ε, φοβάμαι ότι κονδύλια θα δοθούν σε πολυεθνικές εταιρείες ενώ θα έπρεπε μεγαλύτερο ποσοστό των κονδυλίων να εκταμιευτεί σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν μπορούν να λύσουν δάνεια από την αγορά. Ε, Εξάλλου ε, και το ε, Ταμείο της Έρευνας και αυτό θα πρέπει κατά την άποψή μου να χρηματοδοτεί. Ε, και αν δεν διαφωνείτε να πω και τη δική μου, τη, τις δικές μου αφού τέλειωσα με αυτές του συναδέλφου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον Χωσέ Μανώλη και τον Ούντο για τη δουλειά που έκαναν. Είναι σαπές ότι την έχουν ξανακάνει κατά το παρελθόν. Γιατί έχουμε μπροστά μας ε, και γενικώ έχουμε μια πολύ καλή υπεπειραμένη ομάδα. Η έκθεση λοιπόν μας ε, σκιαγραφεί πάρα πολύ καλά το που ακριβώς βρισκόμαστε και που πορευόμεθα. Στα περισσότερα τμήματα της έκθεσης ε, συμφωνώ με τα συμπεράσματά σας. Η επικοινωνία και η μεγαλύτερη διαφάνεια είναι το κλειδί για να είναι το έψη πιο επιτυχημένο ε, το ΕΨΙ έχει πραγματικά ξεπεράσει τις ε, προσδοκίες μας. Πρέπει να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες για να είναι καινοτόμες, να προχωρήσουν τεχνολογικά. Πιστεύω ότι η τεχνολογική πρόοδος ε, θα πρέπει να υπάρχει σε όλες τις περιφέρειες με την ίδια ταχύτητα. Να σας πω επίσης ότι η ε, συμβουλευτική που προσφέρεται δεν τη χάνει πλήρους εκμετάλλευσης. Με καλύτερη επικοινωνία και δουλειά επιτόπου στις περιφέρειες το πρόγραμμα ΕΨΗ μπορεί να αποφέρει πολλά περισσότερα. Η έλλειψη ενημέρωσης ε, απορρέει από πολλά, ίσως ε, διότι είναι ένδειξη καταρχήν ε, του πόσο γρήγορα προχωρά ένα πρόγραμμα. Νομίζω ότι γενικά στην αρχή υπήρχαν κάποια αρνητικά συναισθήματα έναντι της συμβουλευτικής. Μερικοί εξημών κατάλαβαν ότι είναι μια πλατφόρμα, ότι πρέπει να μπούμε σε αυτή την πλατφόρμα και ξαφνικά αν μπούμε θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Αλλά αυτή η προσέγγιση δεν ήταν ιδιαίτερα λειτουργική. Νομίζω πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τις διαφορές ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη και η συμβουλευτική που υπάρχει επιτόπου στις περιφέρειες αυτή μπορεί να είναι πολύ πιο πολύτιμη. Αυτά είχα να σας πω και προσβλέπω σε αγαστή συνεργασία με τον Ούντο και τον Χωσέ Μανουέλ. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή οι δύο σκιώδεις της Γκουε δεν είναι εδώ, ε, ο Ντεμάση, κύριος ε, ε, Νιριάντα, ο κύριος Βιέγκ θα λάβει το λόγο. Καλό σας βράδυ. Πιστεύω ότι αυτή η έκθεση σχετίζεται καταρχήν με το σχέδιο Γιούνκερ και θεωρώ ότι το ΕΦΣΥ δεν ακολουθεί απόλυτα τη λογική του ε, σχεδίου σε σχέση με, τη δημόσια, με τις δημόσιες επενδύσεις και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Δηλαδή, χρειάζονται υποδομές στην Ευρώπη, στις περιφέρειες και ούτω καθεξής. Χρειάζεται λοιπόν ένα δημόσιο σχέδιο επενδύσεων. Εδώ μιλάμε για ιδιωτικές επενδύσεις που δίνουν χώρο στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Δηλαδή χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν της πείνας, αλλά υποτίθεται ότι δεν υπάρχει κάποιο χάσμα ως προς αυτό. Θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση μιλάμε για την εφαρμογή του σχεδίου. Υπάρχουν πολλές επικρίσεις σε σχέση με την επικέντρωση σε τομεί σε ορισμένες χώρες και μέσα στα πλαίσια της προσθετικότητας. Δηλαδή γίνονται επενδύσεις από πλευράς ιδιωτικών επιχειρήσεων και έτσι Θεωρώ ότι το σχέδιο Juncker δεν έχει προβεί σε μία μελέτη αντικτύπου. Είναι πολύ νωρίς για να αποτιμήσουμε το σχέδιο. Φυσικά υπάρχει και έλλειψη σωστής επικοινωνίας. Αλλά θεωρούμε ότι γενικότερα είναι πρόωρο να παραταθεί ένα τέτοιο σχέδιο και εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε την εγγενή λογική του σχεδίου και του ταμείου. Alors, Jordi Sol. Eh Thank you, Chair. Oui. Let me... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να αρχίσω ευχαριστώντας τους εισηγητές για τη δουλειά που έκαναν και να καλωσορίσω ιδιαίτερα τον τόνο αυτής της έκθεσης που ισορροπεί μεταξύ μιας θετικής αξιολόγησης του ΕΦΣΥ ως πρωτοβουλίας δημόσιας για την ε, υποβοήθηση των επενδύσεων και της αυτονομίας των πολιτών και από την άλλη υπάρχει μια ε, επικριτική νότα σε σχέση με τη διαχείριση του Ταμείου μέχρι τώρα. Ο, απότατο ο απότατος στόχος του Ταμείου ως δημόσιο μέσο είναι να κινητοποιήσει στρατηγικές επενδύσεις που θα δημιουργήσουν μακροπρόθεσμα ωφέλη για τους πολίτες της Ένωσης, ποιοτική απασχόληση και μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην ενέργεια, ε, τηλεπικοινωνίες, στην υγεία, την παιδεία, ε, και στον τομέα των υπηρεσιών που είναι σημαντικές ε, στην οικονομία. Ενώ ε, η κινητοποίηση κονδυλίων είναι ένα μέσο, δεν είναι αυτός σκοπός. Το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα είναι σημαντικό για τις επενδύσεις και το απτό οικονομικό όφελος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ίσως πολύ νωρίς ακόμα να πούμε αν είναι αποτελεσματικό εργαλείο το ΕΦΣΙ για να ε, οδηγήσει την οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη. Τα έργα πρέπει να εστιάζουν επίσης σε στρατηγικούς τομείς ε, ευθυγραμμισμένα με την πολιτική της Ένωσης και τα κοινωνικά ωφέλη. Ε, γι' αυτό είμαστε απογοητευμένοι από την υποστήριξη του ΕΦΣΙ στο θέμα των ορυκτών καυσίμων. μόνο ένα τέταρτο των ενεργειακών project ε, ήταν στα ορυκτά καύσιμα. Αυτό είναι επιβεβαιωμένο. Είναι σημαντικό το θέμα των ορυκτών καυσίμων ε, για το μέλλον και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται δημόσια κονδύλια για να ε, υπονομεύονται οι προσπάθειες για το κλίμα σε επικίνδυνες δηλαδή ε, πηγές ενέργειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά το ΕΦΣΥ, μιλήσαμε ενδελεχώς τα τελευταία χρόνια και όσον αφορά τη δική μου ομάδα θέλω να σας πω ότι είναι, είναι ένα πολύ μεγάλο στρατηγικό λάθος διότι η ευρωπαϊκή οικονομία αυτή τη στιγμή ε, διέρχεται μια μεγάλη κρίση ζήτησης και το ΕΦΣΥ ως εργαλείο ε, προσθέτει περισσότερο στη ζήτηση στην προσφορά, με συγχωρείτε, στην προσφορά, όχι στη ζήτηση. Άρα δηλαδή ήδη από τη βάση του δεν καλύπτει τις ανάγκες οικονομίε και αυτά που χρειάζεται η πολιτική στην Ευρώπη. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτή την παραδοχή ε, ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ζήτηση, είναι σαφές ότι θα πρέπει να βρούμε κάποιες άλλες εγγύσει για τις επενδύσεις που θα πρέπει να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αν δεν το κάνουμε αυτό δεν θα προκύψει ουσιαστική προσθέμενη ε, αξία εργασία παρά μόνο περισσότερα χρήματα στα, στις τσέπες πολύ λίγων όπως έχουμε δει ήδη από την εφαρμογή μέχρι τώρα του ΕΦΣΥ. Για την προσθετικότητα συμφωνώ με τους εισηγητές ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται κριτήρια όπως είναι η καινοτομία, η ενεργειακή μετάβαση, τα ορυκτά καύσιμα, η αυτοκινητόδρομη, η υποδομή, όλα αυτά δηλαδή που προσφέρουν προστιθέμενη αξία. Ε, και μέχρι τώρα δεν υλοποιήθηκαν όλα αυτά γιατί Προφανώ ακολουθείται και μια διαφορετική ε, κατεύθυνση. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να επιμείνουμε σε κάτι, να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, γιατί στα 93 προγράμματα που μέχρι τώρα εγκρίθηκαν, ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, στοιχεία που είναι κάπω μπερδεμένα. Εμεί θέλουμε καλύτερε, πιο διαφανεί αξιολογήσει, γιατί πρέπει να γίνονται οι αξιολογήσει και σε εθνικό επίπεδο. Θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογούμε τις επενδύσεις και από άλλες πλευρές, όχι μόνο να περιζόμαστε σε αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ε, ΕΤΕ, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Για από το EFTD δεν υπάρχει κανείς ούτε από την ΕΝΕΦ, e άρα ο Μάρκο Τζάνι έχει το λόγο. Ευχαριστώ. το πιο ουσιώδες πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε στο ΕΦΣΥ ήταν η χρήση αυτής της μόχλευσης και στην ουσία φτάσαν χρήματα στα κράτη-μέλη για ερευνητικά και αναπτυξιακά σχέδια. Η έκθεση που είδαμε και σύμφωνα με τον ε, κανονισμό που προϋπάρχει δεν ήταν πολύ ε, σαφές, δεν ήταν σαφές κατά πόσα αυτά τα χρήματα μπήκαν σε σχέδια που έχουν προσθετικό χαρακτήρα και από αναλύσεις που έγιναν φαίνεται ότι το 90% των σχεδίων που χρηματοδοτήθηκαν είναι σχέδια που δεν είχαν αυτό το χαρακτήρα της ε, προσθετικότητας όπως θα έπρεπε. Και αυτό διείπε και όλη την ιστορία του ΕΦΣΙ Εξ ονόματος της ομάδας μου η αξιολόγηση είναι αρνητική. Θα δούμε ποια θα είναι και τα αποτελέσματα σε σχέση με τη συνεισφορά στην ε, αύξηση του ΑΕΠ, εάν δηλαδή θα υπάρχει ένα ορατό αποτέλεσμα. Εγώ δεν το πιστεύω. Τότε όμως θα κρίνουμε καλύτερα αυτό το σχέδιο. Ο μόνος τρόπος ε, για να προωθηθεί η έρευνα και η ανάπτυξη μέσω επενδύσεων είναι ε, με ένα ευρύ πρόγραμμα ε, δημοσίων επενδύσεων γιατί ο ιδιωτικός τομέας δεν έχει τα ίδια συμφέροντα με το δημόσιο και αυτά τα αποτελέσματα δεν θα είναι καθόλου ικανοποιητικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε καθυστερήσει, λυπάμαι γι' αυτό δεν θα έχουμε catch the eye και δίνω το λόγο στον κύριο Άντζελ στην Επιτροπή για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω όλοι πιστεύουμε ότι το ΕΦΣΙ έχει επιτυχία και ότι το σχέδιο ανταποκρίνεται ίσως ό,τι αφορά φιλοδοξίες και όγκο Εντοπίσαμε και κάποιες αδυναμίες βέβαια που πρέπει από κοινού με το Κοινοβούλιο να ε, αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν πέντε τομείς όπου προτείνουμε να επιφέρουμε σημαντικές βελτιώσεις. Το ένα είναι η προσθετικότητα που είναι δύσκολη ιδέα ε, αφεαυτής είναι δύσκολο να αποδειχθεί ότι υπάρχει. Ήδη επιτύχαμε σημαντική πρόοδο γιατί βοηθήσαμε να επικεντρωθούν σε, πιο, σε, σε μεγαλύτερου ρίσκου ε, δραστηριότητες, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο. Γι' αυτό η Κομισιόν πρότεινε να δημιουργήσει ένα νέο, ε, κάποια καινούργια κριτήρια επιλεξιμότητας, όπου όλα τα έργα θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις, ότι δηλαδή θα πρέπει να αντιμετωπίζουν μια κατάσταση ε, επενδυτική υποβέλτιστη ή κάποιο κατεπήγον ζήτημα. Δεύτερον, μεγαλύτερη διαφάνεια. Πολλές φορές ε, αμφισβητείται το ΕΦΣΙ και ο τίτλος του, καμιά φορά ε, υπάρχει ένα ερωτηματικό σε σχέση με το αν είναι οι κατάλληλες οι υπηρεσίες, αλλά ως επιτοπλίστων ε, η αμφισβήτηση υπάρχει γιατί δεν γνωρίζουν πολλά για το ΕΦΣΥ. Πρέπει λοιπόν να δημοσιεύουμε τους πίνακες επιδόσεων, και οι επενδυτικέ επιτροπέ να κοινοποιούν τις αποφάσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με αιτιολόγηση, δηλαδή αυτό το έργο σέβεται τι προποθέσει διότι α, β, γ, δ. Όλοι λοιπόν να καταλαβαίνουν γιατί ελήφθη η συγκεκριμένη απόφαση και έτσι και ο νομοθέτη, στο Κοινοβούλιο να ε, ε, διασφαλίζει ένα πλαίσιο λογοδοσίας. Ε, γεωγραφική ισορροπία. Η Κομισιόν δεν είναι ικανοποιημένη από την υφιστάμενη γεωγραφική κατανομή στο ΕΕΦΣΗ και θέλουμε να τη βελτιώσουμε βελτιώνοντας ε, το, την πλατφόρμα της συμβουλευτικής ε, να είναι πιο προορατική, να είναι επιτόπου ούτω ώστε το ΕΦΣΙ να φτάσει σε κάποιους τομείς που θα διευκολύνουν έργα σε άλλα κράτη-μέλη. Επίσης χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα για τις ΜΜΕ, αυτό είναι το τέταρτο. Σίγουρα υπήρξε ανταπόκριση, αλλά μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Και τέλος πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επιτελέσουμε πρόοδο στην κλιματική αλλαγή γιατί έχουμε το στόχο να αυτό να ε, βελτιώσουμε την καταπολέμηση της ε, κλιματικής αλλαγής. Σταματώ εδώ. Συμφωνούμε με το Κοινοβούλιο που θέλει να βελτιώσει ε, την προϋπόθεση για τη φορολόγηση. Αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να υπάρχει στο κείμενο και εδώ επιτελεί πρόοδο η Τράπεζα Επενδύσεων. Για τον προϋπολογισμό αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιοι από εσά είστε απρόθυμοι να πάρετε από το μέσο συνδέοντα στην Ευρώπη άλλα χρήματα, αλλά αυτά θα μπορεί να χαθούν γιατί δεν υπάρχει pipeline τώρα. Και για τη διακυβέρνηση είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε επικοδομητικά με το Κοινοβούλιο για να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ευχαριστώ. Τώρα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει το λόγο. Ποιο θα εκφραστεί, ο κύριος Μόλτερερ. Για δύο λεπτά σας παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε πολλοί στην αίθουσα. Θα ήθελα λοιπόν να μην γίνονται συζητήσεις μεταξύ σας για να ακούσουμε τον κύριο Βόλτερερ. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι ε, είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένο με τι συζητήσει που γίνονται στο Κοινοβούλιο, όχι μόνο βέβαια με τι σημερινέ, αλλά αυτή η συζήτηση και η επικοινωνία με το Κοινοβούλιο ήταν και είναι, εξακολουθεί να είναι το κλειδί για την εφαρμογή του ΕΨΗ και θα παραμείνει και το κλειδί, ο καθοριστικό παράγων για το μέλλον. Θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάποια άλλα θέματα που κατά την άποψή μου υπάρχει περιθώριο βελτιώσεων. Η κατανομή των χωρών είναι κάτι που βλέπουμε να υπάρχει περιθώριο ε, βελτιώσεων. Μπορεί λοιπόν να συμβεί το εξή. Ε, Αυτό ο κόμβο συμβουλευτική μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικό τόπου να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητε κάθε περιοχή. Δεύτερον, να υπάρχουν οι πλατφόρμε επενδύσεων και η συνεργασία με τι εθνικέ επενδυτικέ τράπεζε, να βελτιωθεί αυτή η συνεργασία. Και τρίτον, να υπάρχει καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στο ΕΦΣΙ και τα διαρθρωτικά ταμεία. Να συνδυαστούν αυτά τα δύο μέσα. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τον κανονισμό που προβλέπει ε, και άλλους ε, τομείς ε, που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν. Η έκθεση καλύπτει και ένα άλλο θέμα, το υπερεθνικό στοιχείο. Προς το παρόν δεν έχουμε υπερεθνικά προγράμματα ανάμεσα σε περισσότερα κράτη-μέλη και αυτό είναι μια αδυναμία που έχει προκύψει κατά την εφαρμογή. Τέταρτον, χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία για την προσθετικότητα. Αυτό σημαίνει και μεγαλύτερη διαφάνεια. Πολύ σωστά, μερικοί εξημών αναφέρατε ότι ε, ο κανονισμός που υπάρχει είναι και η σωστή κατευθυντήρια γραμμή για το ε, πίνακα επιδόσεων. Και θέλω να σας πω ότι η Επιτροπή που ασχολείται με τις επενδύσεις αποτελεί ιδιαίτερη σημασία στην προσθετικότητα και στον, σκόρο, ε, στον πίνακα επιδόσεων για να αποδείξουμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερες πληροφορίες αλλά και να σας προσφέρουμε και μεγαλύτερη ασφάλεια. Και τέλος θέλω να πω Μακροπρόθεσμα βλέπω ότι υπάρχει και κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Είναι η εξέλιξη των αγορών όσον αφορά στις ρυθμίσεις των αγορών. Μην ξεχνάτε ότι το επενδυτικό πρόγραμμα της Ευρώπης βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Το ΕΦΣΙ είναι το ένα, ο ένας πυλώνας ε, οι κανονισμοί ε, και η συμβουλευτική, αυτά τα τρία αποτελούν, είναι εξίσου σημαντικά όσο και το ΕΦΣΥ. Ευχαριστώ πολύ το Γενικό Διευθυντή. Ε, εντάχει οι δύο μας εισηγητές ένα λεπτό ο καθένας. Θα να σας ευχαριστήσω για την έκθεση που μας υπέβαλαν που είναι πολύ σημαντική για το FC2 που θα είναι η συνέχεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Στην πρώτη του φάση ποιος θα αρχίσει, ο κύριος Μπούλμαν. Αγαπητοί μου συνάδελφοι, σας ευχαριστώ θερμά. Είμαι βέβαιος ότι... Ε, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα αντιμετωπίσουμε με μεγάλη προσοχή οι δύο εισηγητές τα, τις παρατηρήσεις σας. Να σας πω πάλι την προθεσμία κατάθεση στην 28η Φεβρουαρίου. Περιμένω τις τροπολογίες σας. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Αβζελ πολύ, με πολύ ακριβή και σαφή τρόπο ε, τόνισε τα θέματα που πρέπει να βελτιωθούν, να τροποποιηθούν και κατά τη γνώμη της Κομισιόν και πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο παρόμοιες εκτιμήσεις θα κάνει και γι' αυτό θα επεξεργαστούμε επικοδομητικές λύσεις τελικές. Ε, έλαβα υπόψη μου τις παρατηρήσεις του κυρίου Μόλτερ επίσης ότι υπάρχει προθυμία από τους υπεύθυνου στο ΕΦΣΙ ε, για να υποστηρίξουν τις βελτιώσεις όχι τώρα που συζητάμε αλλά και στην πράξη αργότερα για να βελτιωθεί το ΕΦΣΙ 2. Κύριος Φερνάντες, εδώ και ένα μισή χρόνο μιλούσαμε για αυτό το ταμείο με πολλές αμφιβολίες, αν θα μπορούσε να λειτουργήσει, αν θα υπήρχε καν και κατά πόσο θα τηρούνταν οι προδιαγραφές στον τομέα του περιβάλλοντος. Σήμερα μιλάμε για επέκταση του Ταμείου. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ε, επενδύσεις της ΜΜΕ και μιλάμε για 500 δις ευρώ. Το Ταμείο λειτουργεί καλύτερα και μπορεί με τον υπάρχοντα κανονισμό να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα. Θα πρέπει όμως να κάνουμε διευκρινήσεις για τον νέο κανονισμό. Ε, χρειάζονται επενδύσεις ιδιωτικές και δημόσιες. Οι ιδιωτικές επενδύσεις δεν σημαίνει ότι είναι κακές εξορισμού. Μπορούμε να συνδυάσουμε τις δύο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και πολλές δημόσιες επενδύσεις έγιναν από το ΕΦΣΥ. Σε μας δόθηκαν 250 εκατομμύρια ευρώ σε επίπεδο δημοτικών αρχών Λισαβόνας. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλες σας τις παρεμβάσεις και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεισφορά σας σε αυτή την έκθεση εφαρμογής και για την επέκταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Ευχαριστούμε τους εισηγητές. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατί το ξεκίνημα είναι πολύ θετικό, αλλά υπάρχουν και περιθώρια βελτίωσης βασιζόμαστε σε εσά για να ασκήσετε πίεση προς την ΕΤΕ. Σταματάμε λοιπόν εδώ ως προς την έκθεση εφαρμογής του ΕΦΣΙ και από εδώ και στο εξής ο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη θα προεδρεύσει. Ευχαριστώ πολύ Ζαν. Περνάμε στις ψηφοφορίες. Όπως Λ... ξέρετε... Ψηφίζουμε για την ε, Ευρωζώνη και θα ήθελα να σας ζητήσω να ψηφίσουμε ε, δοκιμαστικά για επαλήθευση αν λειτουργούν οι κάρτες. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Still a couple colleagues to vote. Ακόμα πρέπει να ψηφίσουν και κάποιοι συνάδελφοι. Ένας πρέπει ακόμη να ψηφίσει. Πέρασε. Εντάξει. Ε, αρχίζουμε λοιπόν. Συμβιβαστική 1. Α, υπέρ κατά αποχές δεκτή η συμβαστική α. Η συμβαστική D υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τώρα πρέπει να πάμε στη σελίδα 16 του καταλόγου. Είναι πολλές οι σελίδες. Συμβιβαστική, ε, ε τροπολογία 264, συγγνώμη, ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 271 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 307 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 323 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, συμβιβαστική ε υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τώρα πάμε στην 24. Συμβιβαστική F ε υπέρ κατά αποχές δεκτή. 33 σελίδα. Συμβιβαστική G υπέρ κατά αποχές δεκτή. 38 σελίδα 38 συμβιβαστική H υπέρ κατά αποχές δεκτή. Σελίδα 44 η 729 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 732 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική I, Ι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Σελίδα 49 τώρα και η συμβιβαστική C υπέρ κατά αποχές δεκτή 57, σελίδα 57, συμβιβαστική B υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή και τέλος με ονομαστική ψηφοφορία, τελική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Vote is closed. Πέρας της ψηφοφορίας. 54 υπέρ, 28 κατά, 6 αποχές, δεκτή η έκθεση, δε συγχαρητήρια στους εισηγητές. Και τώρα πάμε στην ψηφοφορία έκον. Να δώσουμε... Να να, να, να μιλήσουμε κι εμείς. Ναι, πριν μιλήσετε εσείς, θέλω να πω ότι υπάρχει γνωμή ε, μειοψηφία στη CCR που βεβαίως θα περιληφθεί στα πρακτικά. Και με χαρά δίνω το λόγο στους ε, εισηγητές. Ο κύριος Μπέγκε. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Ξέρετε ότι ένα χρόνο εργαζόμαστε πάνω στην έκθεση αυτή και ότι ήταν αρκετά περίπλοκο το εγχείρημα με πολύ καλή θέληση, με πολλή συμβολή από πολλά μοντέλα και απόψεις για το πρακτέο στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία τώρα παλεύει για την ύπαρξή της. Υπάρχουν διαφορετικές υπόψεις, από απόψεις για το ποιος είναι ο καλύτερος δρόμος. Αυτό ήθιστε στην πολιτική αντιπαράθεση ε, και ε, είναι δεδομένο ε, αφού υπάρχουν διαφορετικά προγράμματα των πολιτικών ομάδων. Η αρχή ήταν δύσκολη, μέσα από πολλές τροπολογίες προσπαθήσαμε να βρούμε ένα νέο σχήμα στην έκθεση, ένα νέο μορφότυπο αν θέλετε, ώστε να αυξήσουμε την συνένεση και να μην εμπλακούμε ε, και χαθούμε σε πολλές συμβιβαστικές και στη συνήθη διαδικασία ε, με τις πολλές συζητήσεις. Τώρα νομίζω ότι τα καταφέραμε. Υπάρχουν πολλοί που ενοχλούνται και εγώ ενοχλούμαι ε, σε κάποια σημεία, αλλά αυτό είναι ο συμβιβασμό. Τώρα νομίζω ότι βρήκαμε ένα δρόμο που θα μας επιτρέψει την πέμπτη σε ένα συνολικότερο πλαίσιο τριών εκθέσεων να δώσουμε τα απαραίτητα πολιτικά μηνύματα σχετικά με το τι αναμένουμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι προοπτικές ε, θέλουμε να συζητηθούν και να αποφασιστούν. Αυτό που μας χωρίζει ακόμα, θα, αν προχωρήσει, θα αποτελέσει κομμάτι της νομοθεσίας. Δηλαδή ε, δεν ε, θα μείνουμε ε, σε αυτά που ψηφίσαμε και στα ψηφίσματα που υπάρχουν. Ε, υπάρχει ανάγκη για πολύ εντατικέ και δύσκολες διαπραγματεύσεις που θα αλλάξουν ορισμένα πράγματα. Μας ενδιαφέρει όμως να συγκεντρώσουμε πλειοψηφία ε, να συμφωνήσουμε παρόλο που μπορεί να διαφωνούν ακόμα ορισμένοι. Να βρούμε έναν ε, τρόπο, να δείξουμε ότι είμαστε διατεθειμένοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προωθήσουμε τα συμφέροντα των πολιτών και των κρατών, το λέω συνειδητά με αυτή τη σειρά, και να συμμετέχουμε σε βαρύνουσες αποφάσεις που ξέρω ότι δεν ε, θα είναι εύκολες και δεν θα μπορούν να δικαιολογηθούν από όλους μας τις χώρες μας. Αλλά η συμβιβαστική λύση πρέπει να βρεθεί η Καγκελάριος ε, στην πρώτη ομιλία το 2007 ο Καγκελάριος είπε ότι η ψυχή της Ευρώπης είναι η ανεκτικότητα. Πρέπει λοιπόν να μπορούμε να βλέπουμε και να μπαίνουμε και στη θέση του άλλου. Αυτή η προσέγγιση προς τους άλλους επιτρέπει να βρεθούν λύσεις ε, και προφανώς ε, θα ε, συνεχίσουμε να δίνουμε μάχες για αυτές. Σήμερα πιστεύω ότι κάναμε ένα βήμα μπροστά. Ευχαριστώ την συνεισηγήτρια και τους συναδέλφους από τις πολιτικές ομάδες που συμφώνησαν στην έκθεση αυτή. Ευχαριστώ θερμά για την πολύ εντατική συνεργασία. Δεν είναι μόνο πνευματική άσκηση αυτό που κάναμε τώρα, αλλά ελπίζω ότι την Πέμπτη, αν εγκριθεί η έκθεση, θα έχει γίνει ένα βήμα μπροστά και σε σχέση με τις λύσεις, αλλά και σε σχέση με την αξιόπιστη εκπροσώπηση ε, και τον προσανατολισμό, το σωστό προσανατολισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ, υπερβάνω Περές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο και εγώ θα μιλήσω ως συνεισηγητρία. Ο κ. Μπέγκε το είπε προηγουμένως ότι εδώ και πάνω από ένα χρόνο έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας. Και τώρα έχουμε την αίσθηση ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί συμβασμό. Μπορώ όμω να διαβεβαιώσω όλου του αδέλφου ότι τα καταφέραμε μια χαρά. Γιατί με τον κύριο Μπέγκε τη εξ αρχή ε, είχαμε την θέληση να συμφωνήσουμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το θέμα. Θα ήθελα επίσης να τον ευχαριστώ θερμά για την ε, για το πολιτικό του θάρρος. Ε, και ούμονον αυτό, νομίζω ότι θα πρέπει να επενέσω και την ε, πνευματική ειλικρίνεια με την οποία χειρίστηκε το θέμα. Βεβαίως δεν έχουμε ακόμα ολοκληρώσει, όλοι θα εξαρτηθούν από την ψηφοφορία την Πέμπτη, αλλά νομίζω ότι κάναμε ένα βήμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Με πάση περιπτώσει είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όχι μόνο κατορθώνει να επιτυγχάνει συμβιβασμούς αλλά και ισορροπίες. Και οι ισορροπίες αυτές επιτρέπουν να αποθέτουν τις ελπίδες τους οι άλλοι θεσμοί σε εμά, οποτεδήποτε είναι απαραίτητο να ταρακουνηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς διακυβεύεται. Με το ψήφισμα αυτό όχι βέβαια, δεν είναι ότι ανοίγουν ότι κλείνουν πόρτες, του αντίον ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο. Ε, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά είχαμε παραδείγματος χάρη ε, πέντε προέδρους ε, που τοποθετήθηκαν και εδώ επιπλέον υπάρχει δυνατότητα, όπως σας είπα, να τρακονηθούν πάρα πολύ αρμόδιοι και να γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι όταν θα εκδώσει, θα κοινοποιήσει την ε, Λευκή της Βίβλου, οφείλει και αυτή να εμπνευστεί από τη δική μας ε, την ισορροπία και τους ε, συμβιβασμούς. Ευχαριστούμε όλους τους σκιώδης όλους όσοι συνεργάστηκαν με ζήλο χωρίς να υπολογίσουν ούτε χρόνο ούτε κόπο για να καταλήξουμε σε αυτό το πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάλι λοιπόν συγχαρητήρια στους εισηγητές και εγώ νομίζω ότι η συνεργασία ανάμεσα στις δύο επιτροπές ήταν περισσότερο απόγαστη. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές, να τους συγχαρώ, γιατί και οι δύο έδειξαν και κατανόηση και θάρρος και νομίζω ότι είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να εκπέμψει ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα που να αφορά στο μέλλον της Ευρωζώνης και του Ευρώ. Μόλις έγινε λόγος για το ΕΦΣΥ, πρέπει λοιπόν να κλείσει αυτό το κενό των επενδύσεων. Και θέλω να πω κάτι, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι πολύ σημαντικό να επανέλθει η εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό νόμισμα, στο ευρώ αν θέλουμε να ε, δημιουργήσουμε κίνητρα για θέσει απασχόληση ε, και για επενδύσει. Ευχαριστώ πολύ του συζητητέ. Εύχομαι τα καλύτερα και ελπίζω η Ολομέλεια να επιβεβαιώσει αυτό το αποτέλεσμα τη ε, ψηφοφορία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον όλους. Λοιπόν, τώρα πάλι δοκιμάζουμε ε, το ηλεκτρονικό σύστημα για να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία της Επιτροπής